είναι η σύντομη παρουσίαση, η έκθεση του Μιχέλ Άγγελ Μαρτίνες. Πρόκειται για την σύσταση που αφορά την καταγγελία 185-2005. 2005, ένας διερμηνέας freelance που συμπλήρωσε τα 65 σταμάτησε πλέον να έχει δουλειά από τις ε, ευρωπαϊκά όργανα και κατέσε μια καταγγελία. Πριν από μερικά χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή είχαν αποφασίσει να μην προσλαμβάνουν διερμηνείς freelance ε, μετά από τα 65 τους. Σε, οι διερμηνείς ε, προσέφηγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κέρδισαν την υπόθεση. Αποφασίστηκε ότι υπήρχε διάκριση και παραβίαση του ε, χάρτη θεμελιωθών δικαιωμάτων και ζητήθηκε από την Επιτροπή να αλλάξει τη στάση της αυτής, αναμάντας υπόψη την πρόφαση του Πρωτοδικείου. Εκόφευσε σε αυτά τα οποία είπε ο διαμεσολαβητής ε, ε, η Επιτροπή το θέμα έφτασε στην Επιτροπή Αναφορών και η Επιτροπή Αναφορών για τρεις λόγους υποστήριξε αυτά τα οποία είχε πει ο Μεσομελαβητής με την ε, απόφαση την οποία έλαβε. Πρώτα απ' όλα, διότι θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί με την συμπεριφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο προσλαμβάνει διερμηνείς freelance που έχουν ξεπεράσει τα 65 χρόνια όταν ε, συντρέχουν λόγοι. Δεύτερον, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ο διαμεσολαβητής ε, είναι ε, απαραίτητος για απαραίτητο να δίνει με εντελώ ανεξάρτητο τρόπο την απόφαση. Επίσης, ελέγχθη ότι στην Εγκρίθηκε ένα ψήφισμα, όπως σας λέω, από την Επιτροπή Αναφορών ομόφωνα για το θέμα αυτό και απαιτεί από την Επιτροπή να μπορέσει να συμμορφωθεί στην απόφαση και στην σύσταση την οποία έκανε ο Διόμεσολαβητής. Το ε, ελέγχθη ότι η απόφαση αυτή είναι μία απόφαση η οποία ε, ελήφθη από ένα διοικητικό όργανο και όχι τίποτα περισσότερο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα πω ότι υπάρχει κάποια πρόβλημα, διότι πάντα εμείς ε, προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε την όλη υπόθεση. Έγιναν κάποιες προσπάθειες να μην φτάσει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια και έγιναν και κάποια σχόλια σύμφωνα με τα οποία ό,τι και να αποφασίσει το Κοινοβούλιο δεν θα δοθεί συνέχεια. Πρέπει να πω ότι το θέμα αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχουν κινήσει οι ίδιοι οι αλλά κάποιοι ε, υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τη θέλησή μας πάντα να συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το θέμα αυτό έξω και ελπίζω ότι η ψηφοφορία αύριο θα αντικατοπτρίζει και την ψηφοφορία που έγινε στην Επιτροπή Αναφορών, δηλαδή θα συμφωνεί με την σύσταση την οποία έκανε ο διαμεσολαβητής και έτσι θα μπορέσουν τα πράγματα ομαλά να λυθούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι καλή την πίστη αποφάσισε και έδρασε η Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες. Δεν προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε καμία αντιπαράθεση, ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η άποψή μας ήταν ότι θα αναγνωριστεί η άποψή μας και η θέση μας από τον διαμεσολαβητή. Όλα αυτά τα χρόνια οι συνθήκες εργασίας για τους ε, διερμηνείς συνεδρίων freelance βασιζόταν στους κανόνες ε, του εσωτερικού κανονισμού. Και εδώ και λίγα χρόνια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών ότι μπορούν να πληρώνουν κοινοτικούς φόρους και όχι εθνικούς φόρους, μπήκαν στην κατηγορία αυτή που διέπει ο κανονισμός του προσωπικού καλύπτονται λοιπόν από το άρθρο 19 του κανονισμού των υπαλλήλων και ακριβώς γι' αυτό σήμερα ονομάζονται AIC. Το όριο λοιπόν της ηλικίας των 65 ετών βασίζεται ακριβώς στο όριο όπως ε, για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες υπαλλήλων όλων των κατηγοριών και βάσει του νέου κανονισμού αυτός ο κανόνας ισχύει και εφαρμόζεται και για τους διερμηνείς συνεδρίων freelance το 2000 και το 2004. Μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 2004, όσον αφορά την πρόσληψη διερμηνέων άνω των 65 ετών και την ύπαρξη διακρίσεων βάσει αυτού του κανόνα, το ε, δικαστήριο δημιούργησε μια νέα κατάσταση. Η πρακτική της Επιτροπής μας οδήγησε στην ερμηνεία ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόσει τον κανόνα του Συμβουλίου και να μην προσλαμβάνει άτομα πάνω των 65 ετών, όπως ακριβώς ισχύει για και τις υπόλοιπες κατηγορίες υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες διερμηνίας προσλαμβάνουν τους διερμηνείς βάσει των αναγκών τους, βάσει των αναγκών που ορίζουν οι ίδιες οι υπηρεσίες και εκτιμούν οι υπηρεσίες διερμηνίας. Οι πρώτες ανάγκες αυτών των υπηρεσιών καλύπτονται από υπάλληλους διερμηνείς και οι υπόλοιπε από τις προσλήψεις ε, διερμηνέων freelance, AICs. Από εκεί και πέρα καλύπτονται οι ανάγκες των υπηρεσιών για διερμηνείς και πρέπει να σας πω ότι η πρόσφατη διεύρυνση οδήγησε σε νέες ανάγκες καθώς και την ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των δαπανών. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω την πολύ επικοδομητική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες ο οποίος είχε πολύ καλές και επικοδομητικές επαφές για το θέμα αυτό με τις υπηρεσίες μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες, ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο. Έχετε το λόγο, κύριε Μαρτίνες. Ε, ε, κύριε Πρόεδρε, Έχω ένα λεπτό ακόμη στη διαθέσή μου και θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Επίτροπο που ξέρει πόσο φιλικά διάκυμε και πόσο επίσης φιλικά και του κυρίου Όρμπαν. Δεν είπε τίποτα η κυρία Επίτροπος για την σύσταση του διαμεσολαβητή. Δηλαδή ο διαμεσολαβητής που γνωρίζει όλα τα επιχειρήματα που μας παρουσίασε η κυρία Επίτροπος έκανε μία συγκεκριμένη σύσταση την οποία φαίνεται ότι αγνοεί η Επιτροπή πλήρως. Δεν θέλω να απαντήσει η κυρία Κούνεβα, διότι προφανώς δεν έχει τα στοιχεία εκείνη. Όλα τα στοιχεία που μου έδωσε συμφωνώ με, αυτό το, ε, αυτά τα οποία ξέραμε και αυτά τα οποία ξέρει και ο ίδιος ο διαμεσολαβητής. Δεν μας λέει όμως αν όντως παρόλα αυτά και επειδή ο διαμεσολαβητής γνωρίζει την κατάσταση συστήνει να αλλάξουν οι κανόνες, δεν μας λέει κύριε Επίτροπες, εάν θα ακολουθήσει αυτά τα οποία λέγει ο διαμεσολαβητής και συστήνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την σύσταση που έκανε ο διαμεσολαβητής. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι, νομίζω ότι το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι φυσικά θα επανέλθω, θα ενημερώσω τον Επίτροπο Όρμπαν και είμαι σίγουρη ότι θα έχετε την πρέπουσα απάντηση. Λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη την παρέμβασή σας, καθώς και τα τελευταία στοιχεία διευκρίνησης που μου ζητήσατε. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ την Επίτροπο, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. Τέλος της συνεδρίασης.